Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι εμπειρογνώμονες ε, για την ε, ακρόαση, αλλά έχουμε και τις ε, δικές μας εργασίες για την έναρξη της συνεδρίασης. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω όσους είναι παρόντες και όσους μας παρακολουθούν, διότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή συνεδρίαση. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ηχογραφούνται οι παρεμβάσεις σας. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουν όχι μόνο οι Ευρωβουλευτέ, αλλά και οι εμπειρογνώμονε. Να ξεκινήσω από το πρώτο θέμα τη ημερησία διάταξη, που είναι η έγκριση τη ημερησία διάταξη, η οποία διανομήθηκε στι 7 Ιουνίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή αιτήματα τροποποίησης θα ήθελα να θεωρίσουμε ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Προχωρώ στο τροποποιηση θα μακρηγορήσω ημερησια διαταξη οπω τροποποιηθηκε προχωρω στο δευτερο θεμα τη ημερησια διάταξη οπου θα μακρηγορησω λιγο εχω αρκετέ ανακοινώσεις. Θα ήθελα να σας ενημερώσω καταρχάς ε, ότι όσον αφορά την γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ για τον προϋπολογισμό του 2017 έχουμε νέο χρονοδιάγραμμα το οποίο προτάθηκε από το Κοινοβούλιο λόγω της ε, καθυστερημένης υιοθέτηση από την Επιτροπή του Σχεδίου Προϋπολογισμού για το 2017. Αυτό σημαίνει ότι η παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, και των τροπολογιών που θα γίνουν μόνο στα αγγλικά από τον εισηγητή θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου και αυτό θα γίνει παρουσία του Γενικού Εισηγητή Jens Γκάιερ. Η τροπολογία για την υποβολή τροπολογιών στα αγγλικά αποκλειστικά θα είναι 19 Ιουλίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην ΑΦΚΟ θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου. Θα ενημερωθείτε γραπτός σχετικά με την ε, τροποποίηση αυτή του χρονοδιαγράμματος. Δεύτερον, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες ε, της ομάδας εργασίας ε, για την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία συνεργαζόμαστε στο θέμα αυτό με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων σύμφωνα με τον ε, κανόνα 55. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Μπούζεκ και τον Ράινερ Βίλαντ ως πρόεδρο της ομάδας εργασίας για τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου. Μέχρι στιγμής έχουμε συζητήσει ότι για την ΑΦΚΟ είναι σημαντικός ο προγραμματισμός καθώς και η επαλήθευση της νομικής βάσης καθώς και οι πιθανές ε, τροποποιήσεις της ε, νέας ε, διαθεσμικής συμφωνίας, διοργανικής συμφωνίας. Και επίσης, όσον αφορά την καλύτερη νομοθεσία, θα θυμάστε ότι ο κύριος Σούλς, πρόεδρος του Κοινοβουλίου, σε ομάδα υπό την ε, προεδρία του κυρίου Φερχόφστατ και με ε, παρουσία των προέδρων ε, της ΑΦΚΟ και της Ιούρι καθώς και των δύο επιτροπών για την ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας πρότειναν να υπάρξει άμεση συνέχεια στις εργασίες της συμφωνίας και υπέβαλαν προτάσεις σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτό θα αποφασιστεί από τη διάσκεψη των Προέδρων. Ε, συμμετέχουν ε, λοιπόν όχι μόνο οι διάφορες επιτροπές, αλλά και η διάσκεψη των Προέδρων, καθώς και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Αποφασίστηκε κατόπιν ε, πρότασης της ομάδας αυτής όπου συμμετείχα και εγώ Όσον αφορά τι ε, διαπραγματεύσει για διεθνεί συμφωνίε από πλευρά του Κοινοβουλίου, ο Μπέντ Λάνιε ω πρόεδρο ε, τη ΙΝΤΑ και ο Έλμαρ Μπρόκ ω πρόεδρο τη ΑΦΕΤ να συμμετέχουν. Η ομάδα εργασία ε, που δημιουργήσαμε όμω θα είναι η πλατφόρμα όπου θα γίνεται διαβούλευση όλων των επιτροπών και θα γίνονται οι συζητήσει και οι διαπραγματεύσεις ε, για την παρακολούθηση της ε, διοργανικής ε, συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία έχει να κάνει με θέσπιση των κριτηρίων για τις κατεξιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Και εδώ η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων είναι ότι ο Γιώζεφ Σάιερ από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μαζί με τον Ρίτσαρντ Κόρπετ από την Επιτροπή μας, από την ΑΦΚΟ, θα είναι αρμόδιοι για τις διαπραγματεύσεις. Η εντολή θα είναι το ψήφισμα της έκθεσης ΣΑΙΕΡ του 2014 που υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο σχετικά με την ε, ανάθεση ε, νομοθετικών αρμοδιοτήτων. Ε, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σχετικά και με την προσαρμογή του συστήματος προγραμματισμού για την χρονιά αυτή, <clears throat> για την διοργανική συμφωνία. Επίσης, ελήφθη η συμφωνία σχετικά με το πώς ε, θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ε, διαδικασίας αυτής ε, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Και επίσης σεβόμενοι τις εργασίες των επιτροπών που εξετάζουν τις νομοθετικές προτάσεις αποφασίστηκε επίσης ότι σχετικά με την παρακολούθηση τη συνέχεια που θα δίνεται δηλαδή, η παρακολούθηση της εφαρμογής της νέας συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί από τις επιτροπές και από ε, την ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, ε, αλλά και επίσης η διάσκεψη των Προέδρων θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής της έκθεσης αυτής. Αυτά από μένα όσον αφορά τις ανακοινώσεις και το σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θα ήθελα να προχωρήσουμε στην ακρόαση. Να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονες Και όπως γνωρίζετε, η ακρόαση αυτή έχει να κάνει με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς, ε, με ιδιαίτερο επίκεντρο τους... τα Ηνωμένα Έθνη. Η ΑΦΚΟ έχει οργανώσει αυτή την ε, ακρόαση σε συνεργασία με την ΑΦΕΤ. Και οι δύο επιτροπές αυτές λοιπόν έχουν προσκαλέσει τους εμπειρογνώμονε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι έχουμε τρεις εμπειρογνώμονε. Μία τροποποίηση έχουμε στο πρόγραμμα. Η κυρία Λότε Κνούσεν από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, δεν μπόρεσε να έρθει και έχει αντεκατασταθεί από τον κύριο Γιώνας Ιόνσον. Επίσης, ε, ο καθηγητής Γιάνν Ούτερς ε, προτάθηκε από το ΕΛΚ και την ΑΦΚΟ. Επίσης θα έρθει ο κύριος Ματέος Ιρμίνσκι που προτάθηκε από το ECR ε, από την Πολωνία και αντί για την κυρία Λότε Κνούτσον, όπως σας είπα, θα μιλήσει ο κύριος Γιώνας Γιόνσον που είναι αρμόδιος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, παγκόσμια και πολυμερή ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και δεκαετίες ε, συζητάμε πώς μπορούμε να θεσμοθετήσουμε καλύτερα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διεθνείς οργανισμούς. η κατάσταση αλλάζει και έχουμε τώρα την δυνατότητα να είμαστε πλήρες μέλος διεθνών οργανισμών. Το Κοινοβούλιο έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα την αποφασιστικότητά του να βελτιώσει την παγκόσμια διακυβέρνηση και πάντα επισημέναμε την ε, ανάγκη για βελτίωση της ε, παγκόσμιας διακυβέρνησης ε, και στη σημερινή ακρόαση θα επικεντρωθούμε στις πολλές κρίσεις που σχετίζονται με την λειτουργία των διεθνών οργανισμών. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται περισσότερη προληπτική πολυμερής δράση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτή την ισχυρή έκκληση. Έχει τροποποιηθεί η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και έτσι υπάρχουν πολλοί λόγοι για την σημερινή ακρόαση. Δεν θα περιμένουμε άλλο τον ε, πρόεδρο Μπροκ. Ε, θα ξεκινήσουμε την ακρόαση και θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτο στον, στον καθηγητή Γιάνν Βόουτερς που είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών καθώς και διευθυντή του κέντρου του ΛΕΒΕΝ ε, για ε, τις σπουδές παγκόσμιας Κυβέρνησης καθώς και του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου του ε, Καθολικού Πανεπιστημίου του ΛΕΒΕΝ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ο τίτλο τη ε, συγκεκριμένη μου είναι κάπω προκλητικό. Λέγεται Οι Βρυξέλλε συναντούν την Βεσφαλία. Η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΗΕ και σε άλλου ε, διεθνεί οργανισμού. Στι 6 ε, Ιουνίου του 2016, την περισμένη Δευτέρα, η υπάτη πρόσωπο η κυρία Μογκερίνη απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας στα πλαίσια της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη και είπε επιλέξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει στις ε, πολυμερείς σχέσεις και πιστεύει στα Ηνωμένα Έθνη και ότι ε, οι πολυμερείς σχέσεις ε, είναι μια βασική αρχή και προτεραιότητα για την καινούργια παγκόσμια στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Αυτό επιβεβαιώνει το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη στην αποτελεσματική πολυμερή στρατηγική όπως ε, αποτυπώθηκε το 2003 στη σχετική στρατηγική και από τις απαρχές της η Ευρωπαϊκή Ένωση προτιμά αυτήν ε, την διακυβέρνηση, την πολυμερή δηλαδή. Και σε αυτή τη στρατηγική του 2003 ε, υιοθετήθηκε η έννοια της αποτελεσματικής πολυμερούς στρατηγικής Ω βασικό άξονα για εξωτερική δράση. Επίση, η στρατηγική ασφαλείας τονίζει το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών. Οπότε αυτή η άποψη και δέσμευση επιβεβαιώθηκε στην ε, έκθεση του 2008 όσον αφορά την στρατηγική ασφαλεία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης δεσμεύθηκε για το ότι θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολυμερή διακυβέρνηση. Το 2009 τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, οπότε επιβεβαιώθηκε και πάλι αυτή η αρχή και τουλάχιστον 8 φορές ε, αναφέρθηκε η συνεργασία με τον ΟΗΕ ε, και ε, θεωρήθηκε πλέον ότι ρητός η Ευρωπαϊκή Ένωση προσιλώνεται στην συνεργασία με τον ΟΗΕ για αυτή την πολυμερή μέθοδο συνεργασίας. Πάντως, ε, η συνεργασία με τον ΟΗΕ έχει σημαδευτεί και από πολλές δυσκολίες. Πρόκειται για περιφερειακή διεθνή οργάνωση με υπερεθνικά χαρακτηριστικά και έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές προκλήσεις για μια πολυμερή διπλωματία και μιλούμε επίσης για ε, ένα θεσμικό όργανο που έχει ως επίκεντρο ε, τα κράτη-μέλη γι' αυτό και έδωσε αυτό τον τίτλο στην εισήγησή μου. Επίσης πρόκειται και για ένα τίτλο βιβλίου που έχω συγγράψει και πρόκειται να δώσω σε όλους τους βουλευτές ένα αντίγραφο. Οπότε πρόκειται για ένα φόρουμ επίκεντρο τα κράτη-μέλη και επομένως ε, το θέμα είναι ότι έτσι αναδύονται κάποια δικαιώματα συμμετοχής σε διάφορους φορείς του ΟΗΕ. Και επομένως απαιτείται μια επένδυση σε πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο. Και επομένως κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε ε, μια μόχλευση οικονομική και πολιτική. Όμως παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να αποκτήσει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΟΗΕ. Τώρα να δούμε λίγο πώς έχει αυτό το πλαίσιο ε, της ε, ένταξης των ενεργειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του ΟΗΕ. Στη συνέχεια να δούμε επίσης ε, το λειτουργικό μέρος των σχέσεων με τον ΟΗΕ και να δούμε επίσης ποιες είναι οι ευκαιρίες, ποιες είναι οι προκλήσεις. Mm. Πάντως, για λόγους περιορισμένο χρόνο που έχουμε στην ε, διάθεσή μας ασχολούμεθα μόνο με τον ΟΗΕ, υπάρχουν και άλλα διεθνή θεσμικά όργανα και δυστυχώς ε, πολλά από αυτά τα διεθνή όργανα έχουν ως επίκεντρο τα κράτη-μέλη, όπως και ο ΟΗΕ. Επομένως δεν ισχύουν αυτά που λέμε μόνο για τον ΟΗΕ, αλλά και για όλα τα διεθνή θεσμικά όργανα. Και υπάρχουν βέβαια και ε, κάποιες εξαιρέσεις όπως ο ΠΟΕ, όπου είναι πλήρως, πλήρες μέλος ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τα 28 κράτη-μέλη, και η φωνή των 28 ακούγεται διαμέσου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε το G20, το οποίο επίσης δεν ε, έχει επίσημη δομή αλλά και έχουμε τα τέσσερα κράτη-μέλη και επίσης αποτελεί τακτικό μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε αυτή και έχουμε και κάποια άλλα διεθνή όργανα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και επίσης έχει πετύχει ε, να διαδεχθεί τη θέση των κρατών μελών όπως οι περιφερειακοί οργανισμοί για την αλία. Τέλος πάντων δεν μπορούμε εδώ να επεκταθούμε γιατί πιεζόμαστε από το χρόνο. Πάντως υπάρχουν κάποιες ε, δυσκολίες που θα σας αναφέρω. Και οι δυσκολίες που συναντούμε στα πλαίσια του ΟΗΕ ισχύουν και για τις άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς. Για να δούμε πώς έχει το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον ΟΗΕ. Όπως είπα, ότι παραμένει επίκεντρο του θεσμικού αυτού οργάνου το κράτος μέλος. Κοιτάξτε τι λέει στο άρθρο 4 του καταστατικού. Είναι σαφές ότι το κατόφλι εδώ είναι χαμηλό το ΣΥΠΗΝ και λέει ότι κάθε ειρηνικό κράτος μπορεί να γίνει μέλος. Γι' αυτό και έχουμε 193 κράτη-μέλη. Βέβαια, για να είναι κανείς ε, ε, μέλος εκτός από ειρηνικό κράτος πρέπει να είναι κράτος έθνος, όπως αναφέρεται. Και αυτό ισχύει για τους περισσότερους οργανισμούς του ΟΗΕ, αυτές τις ε, εξειδικευμένες υπηρεσίες και υπάρχουν πάρα πολύ λίγες υπηρεσίες του ΟΗΕ που επιτρέπουν ε, σε άλλες, άλλους οργανισμούς να γίνουν ε, μέλη ως οργανισμοί. Είναι ο ΦΑΟ και η Επιτροπή για τον Διατροφικό Κώδικα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να έχει πρωτογνωστικό ρόλο σε αυτούς τους οργανισμούς και θα μπορούσαμε να γυρίσουμε 15 χρόνια στο παρελθόν διότι τότε είπαμε ότι θεωρήθηκε ως ε, στόχος να γίνει πλήρες μέλος το οποίο φυσικά το πέτυχε αλλά δεν ξέρω αν ε, υπάρχει το ίδιο πνεύμα το, το φιλόδοξο όπως τότε αν υπάρχει και τώρα και στους περισσότερους φορείς του ΟΗΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρατηρητής δεν είναι τόσο σπουδαίος αυτός ο ρόλος είναι τόσο παρατηρητής μπορεί να παραστεί σε επίσημες συνεδριάσεις μπορεί κανείς να λάβει το λόγο αλλά για περιορισμένο χρόνο ε, και αυτό αφορά τα κράτη-μέλη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και δεν μπορούν πάντα να ψηφίζουν να λάβουν το, το λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή να προτείνει άλλου για μέλη. Βλέπετε δηλαδή επομένως, ότι δεν είναι τόσο σπουδαίο το να καλέ παρατηρητή. Και μπορεί κανεί να λάβει το λόγο μόνο αφού έλαβαν το λόγο όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Ε, και όπω είπαμε, για μικρότερο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό είναι ένα δικαίωμα συμμετοχή περιορισμένο. Και αυτό ε, μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα η οποία είναι επιδιώξιμη από τα κράτη-μέλη. Επίσης ε, η συμμετοχή μόνος είναι κολοβωμένη και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει να αναβαθμίσει το, το, το, ρόλο της και να γίνει ε, είτε τακτικό πλήρες μέλος είτε να αναβαθμίσει το καθεστώς του διέπει και να γίνει από παρατηρητής να γίνει παρατηρητής με ειδικά ευξημένα δικαιώματα. Όμως και αυτό απαιτήχθη δύσκολο αυτή η προσπάθεια αναβάθμιση. Επομένως, αυτό φάνηκε την περίοδο 2009-2011. Οπότε και απέσπασε περισσότερα δικαιώματα Ευρωπαϊκή Ένωση στην Γενική Συνέλευση. Επρόκειτο για ένα εγχείρημα δύσκολο. Σε διάφορου οργανισμού του ΟΗΕ δεν εκπροσωπείται καν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι καν παρατηρητή. Α πούμε το Συμβούλιο Ασφαλεία. Βεβαίω, στο καταστατικό, στη συνθήκη, διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν να προσκληθεί η πάτη εκπρόσωπο για να προσφέρει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν κατοχυρώνεται θεσμικά. Το πράγματα είναι χειρότερα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως γνωρίζετε, είναι ένας από τους 20 εξειδικευμένου φορείς του ΟΗΕ και παρά το ότι έχει πάρα πολύ σημαντικές ε, ε, αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί επίσης δεν έχει κάποιο θεσμοθετημένο επίσημο ρόλο. Πέρσι τον Οκτώβριο υπήρξε κάποια πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου, ούτω ώστε κάποια στιγμή να υπάρξει ε, εκπροσώπηση της Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Ίσως γνωρίζετε ότι έχουμε το άρθρο 138 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό προκύπτει της Συνθήκης Λισαβόνας Οπότε βλέπουμε ότι για κάποιες ε, αποκλειστικές αρμοδιότητες όπως η νομισματική πολιτική δεν υπάρχει εκπροσώπηση της ε, Ευρωζώνης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ξέρουμε, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την διεθνή εκπροσώπηση. Και σύμφωνα με το άρθρο 17 τη Συνθήκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στα διεθνή φόρα, εκτό από ε, την εξωτερική πολιτική, συγγνώμη, εκτός από την ε, ΔΑΣΕ και είπαμε ότι υπάρχει αυτή η εκπροσώπηση σε υπουργικό επίπεδο. Και σας παραπέμπω σχετικά και στο 16 της Συνήθειας της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τότε που τέθηκε σε η ισχύ τη Συνήθεια Λισαβόνα έχουμε τι αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που ήταν πολύ πετυχημένη η ρύθμιση τη συνθήκη και έχουμε πάνω από 140 τέτοιε πρεσβείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση παντού στον κόσμο. Αλλά έχουμε και τι αντιπροσωπείε ε, και στον ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, στην ε, Γενέβη, σε Παρίσι, Ναϊρόμπι, Βιέννη και Ρώμη. Οπότε βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθημερινά εκπροσωπείται από τις ε, αντιπροσωπίες. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία που επέτυχε, που, τόσο που, που υλοποίησε και τις Λισαβόνας. Τώρα ε, θα πρέπει να υπάρξει κάποιο συντονισμός, ο ώστε να προβάλλει τις θέσεις του. Οπότε εσωτερικό συντονισμός χρειάζεται, ούτω ώστε να ακούγεται ενιαία η φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει συνέπεια στις ψηφοφορίε. Ε, μην ξεχνούμε ότι έχουμε 28 κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη ε, έχουν ευθυγραμμιστεί με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια είναι μια διαδικασία περίπλοκη και μετά τη θέση τη της συνθήκης της Λισαβόνας ε, γίνεται συνεχής προσπάθεια για τον καλύτερο συντονισμό στις ε, Βρυξέλλες ε, με τις ομάδες εργασίας αλλά και επιτόπου ε, στις έδρες των διεθνών θεσμικών οργάνων που έχουμε στις αντιπροσωπείες. Οπότε είναι χρονοβόρα διαδικασία, είναι περίπλοκη ο συντονισμός. Δύσκολο και τα 28 κράτη-μέλη να μπορούν να ευθυγραμμιστούν και να μιλούν με ενιαία φωνή. Οπότε ε, έχουμε επενδύσει σε αυτό και Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κάποιο είδους ε, συνεργασία σε όλες τις περιοχές του κόσμου ε, και κυρίως για τον ΟΗΕ που έχουμε τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα 193 του ΟΗΕ και φυσικά είμαστε εκεί μειοψηφία. Να σας πω λίγα λόγια τώρα για την λειτουργική συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Εθνών, επιτόπου on the ground δηλαδή. Η συνθήκη της Λισαβόνα αναφέρεται σε ορισμένα σημεία σχετικά με τη συνεργασία με, τη, με τα Ενωμένα Έθνη, όπως για παράδειγμα στο κεφάλαιο για την ανθρωπιστική βοήθεια, για την πρόληψη συγκρούσεων κλπ. Στο επιχειρησιακό επίπεδο υπάρχουν σημαντικά βήματα πρόοδου. Μπορεί να πει κανεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως όταν πρόκειται για αναπτυξιακή βοήθεια βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρωτοπορία μεταξύ των ε, παγκοσμίων δωρητών. Πάνω από 50% της συνολικής <clears throat> επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Μέρος των ε, πόρων αυτών, των κονδυλίων αυτών, ε, διοχετεύεται διά των οργάνων των Ενωμένων Εθνών. Πρώτα UNDP, United Nations Development Program, αλλά και FAO, δηλαδή <clears throat> ο οργανισμός ε, αγρο, ε, αγροτικής οικονομίας, γεωργίας δηλαδή και τροφίμων. Και με μεγάλες δημοσιονομικές ας πούμε δωρεές που γίνονται με εθελοντικές δωρεές προς τον FAO και που εν τέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πάνω από 150 προγράμματα του FAO παγκοσμίω. Και βεβαίω η EuroPaid και όσο γνωρίζετε υπάρχει και μια παράδοση αναέτος το FAO Brussels Office εκδίδει εκείνη η έκθεση με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο στην ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και σε ειρηνιστικές αποστολές ή πρόληψη των συγκρούσεων. Τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε δει πολύ σημαντικές συνεργασίες. Το 2003 είχαμε μάλιστα και κοινή διακήρυξη για συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Εκεί υπάρχει και Διευθυντική Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμμετάσχει και στην ουσία σε πολλές ε, αστυνομικές αποστολές διατηρώντας κυρίως την γεωγραφική στόχευση στην Ευρώπη και στην Αφρική. Οι 28 χώρες μέλη συμβάλλουν σε πάνω από τα 2 τρίτα συνολικά του προϋπολογισμού των αποστολών των Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα στρατιωτικό, προσωπικό αλλά και αστυνομικό και παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται μόλις το 5% του συνόλου των παρατηρητών των Ηνωμένων ε, Εθνών. Άρα υπάρχει εδώ μια έλλειψη ισορροπίας. Υπάρχει βέβαια χώρος βελτιώσεως και ιδίως ό,τι αφορά τον σχεδιασμό των εντολών, την εκπαίδευση και την συμβολή των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Και οι δύο αυτοί οργανισμοί, δηλαδή Ένωμενα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν βήματα για να βελτιώσουν το αποτέλεσμα της συνεργασίας, όμως έχουν αναπτύξει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία που οδήγησε τον γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται μαζί στις Βρυξέλλες, να δηλώσει ότι πρόκειται για μια εποχή της συνεργασίας για την ειρήνη. Ας έρθω σε ορισμένα ε, τελευταία τώρα. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, διαρρύθμισε διαφορετικά την αρχιτεκτονική των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τονίσει το στοιχείο της συνέχειας, εξακολουθεί να υπάρχει το δυναμικό το οποίο δεν έχει εξαντληθεί ακόμη για περαιτέρω αύξηση της αποτελεσματικότητας και της σύνοχης της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο πλαίσιο των Ενωμένων Εθνών και μάλιστα και η θέσπιση του λειτουργήματος του αξιώματο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και της εκπροσώπου έχουν συμβάλει πολύ μεγάλα, ε, πολύ ε, σημαντικά μάλλον ε, στην διαμόρφωση των σχέσεων αυτών και επιτρέπουν την δημιουργία μιας θεσμικής μνήμης στην οποία βασίζεται και μια συναγωγή συμπερασμάτων και διδαγμάτων και αποτελεί και υπόδειγμα προς τρίτες ε, χώρες και τα λοιπά. Και θυμηθείτε και την δήλωση παλαιότερα του Χένρι Κίσιγκερ σχετικά με το ποιον μπορώ να πάρω τηλέφωνο στην Ευρώπη για να συνεννοηθώ μαζί του. Ε, υπάρχουν λοιπόν και τα επιτελεία στη Νέα Υόρκη, στην Βιέννη, στην ε, Γενέβη κλπ. που έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και για τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των χωρών μελών επιτόπου αλλά και για να συνεργαστούν και με άλλες χώρες των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να δημιουργηθούν ευρύτεροι συνασπισμοί. Αυτό, όλα αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Βεβαίω, ο συντονισμό έχει βελτιωθεί, ε, γίνεται και καλύτερο σταδιακό και σχεδιασμό των δράσεων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στα διάφορα φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζω επίση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στα Ηνωμένα Έθνη. Πρόκειται για τον πιο επιτυχημένο πολυμερή οργανισμό παγκοσμίω. Και αυτό αποτελεί ένα πραγματικό ε, σημαντικό θετικό στοιχείο για τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτή η συνδυασμένη δύναμη και τα δίκτυα των 28 χωρών μελών μπορούν πράγματι να προσφέρουν ε, πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, ικανότητες, να συμβάλλουν λοιπόν στην διατήρηση της ειρήνης, στην σταθερότητα, και να συνεχίσουν να δίνουν το παράδειγμα ότι η περιφερειακή ενοποίηση αποτελεί μια καλή συνταγή και ότι είναι ακόμη ένα θαυμάσιο εγχείρημα το οποίο επιτρέπει ε, να ελπίζει κανείς ότι θα υπάρξει ε, και μια, ένα πέρασμα από τη περιφερειακή ενοποίηση στην παγκόσμια ενοποίηση. Ωστόσο δεν έχει ακόμα υλοποιήσει πλήρως το δυναμικό της. Το να μιλούν οι χώρες μέλη με μια φωνή δεν φτάνει συχνά δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταφράσει την εσωτερική της συνοχή σε μια φωνή πραγματικής βαρύτητας. Όπως είπα, είμαστε 28 χώρες από 193 στα Ενωμένα ΕΕ Έθνη και επομένως συχνά βρισκόμαστε σε αριθμητική μειοψηφία. Χρειάζεται λοιπόν διαρκώς να γίνεται προσπάθεια για να δημιουργούνται συνασπισμοί διαπεριφερειακή συνασπισμή και έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και γίνεται μάλιστα τώρα και πολύ συστηματικότερα από ό,τι στο παρελθόν. Όμως, όπως είπα, η διαδικασία εσωτερικού συντονισμού μεταξύ 28 χωρών μελών που βασίζεται πάντοτε στη συνένεση είναι δαπανήρης ό,τι αφορά το χρόνο και τους πόρους. Υπάρχει και αυτή η εξωτερική αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενός είδους μπλοκ συνασπισμού όπου ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη όταν μιλούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανακοινοθέντα τους λένε the block <clears throat> σαν να είναι κάτι το άκαμπτο καταλήγουν βεβαίως να θέτουν να προωθούν το μήνυμά τους 28 με κάπως άκαμπτο τρόπο αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα γνωρίζει αυτά και είμαι βέβαιος ότι αναζητεί ρεαλιστικές από δυτικέ λύσει. Υπάρχει και εσωτερική πρόκληση. Δεν έχουμε μόνο δυσκολίε στα Ηνωμένα Έθνη επειδή είναι ο οργανισμός που βασίζεται στο κράτος έθνο. Έχουμε προβλήματα και μεταξύ των χωρών μελών μα, διότι υπάρχει ένας υποβόσκον φόβο της σταδιακής απώλειας κυριαρχίας που κάποια φορά κάνει τις χώρες μέλη να διστάζουν να ενισχύσουν την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη ως συνόλου. Άρα πρέπει πρώτα να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας, εάν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη στρατηγική αποτελεσματικότητα μέσα στα φόρουμ των διεθνών οργανισμών. Και βεβαίως μετά θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε και την υποστήριξη και τρίτων χωρών και του ίδιου του οργανισμού. Κάποιες τρίτες χώρες, μην το λησμονείτε, προτιμούν να βλέπουν διαιρεμένες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει πάντως αυτός ο κίνδυνος. Έχει καλώς. Νομίζω ότι θα ε, αρκεστώ σε αυτά. Κάτι που είναι ακόμη σημαντικό νομίζω είναι αν εξετάσουμε τα περασμένα 10-15 χρόνια η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ ενός μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσεγγίσεως βρήκε απήχηση στα Ηνωμένα Έθνη. Αναπτυξιακή βοήθεια, ανθρωπιστική βοήθεια είναι από τους τομείς όπου έχει αναπτυχθεί η συνεργασία Ενωμένων Εθνών Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στενή και σταθερή συνεργασία, συμμαχία με κοινούς στόχους. Έχουν όμως χαθεί και κάποια πράγματα λόγω των διαφορών μεταξύ του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του θεσμικού πλαισίου των Ενωμένων Εθνών και λόγω φόβων και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από την πλευρά τρίτων χωρών σχετικά με την απώλεια ε, κύρους, με την απώλεια κυριαρχίας και ούτω καθεξής. Τα γνωρίζουν αυτά βεβαίω οι θύνοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν κάποιες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και με αυτά τα λόγια άρχισα και όλα στην ομιλία μου και έτσι θα την τελειώσω, η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των ΗΠΑ και υπέρ της πολυμερούς προσεγγίσεως μένει και θα παραμένει και πρέπει να παραμείνει έτσι. Αυτά είπε και η υπατή εκπρόσωπος την προηγούμενη εβδομάδα. Και η συνολική στρατηγική δείχνει την στάση αυτή. Και όπως είπε η κυρία Μογκερίνη την προηγούμενη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, η δική μας Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανέρχεται πάντοτε στα Ενωμένα Έθνη, στον πυρήνα του Διεθνούς Πολυμερούς Συστήματος και στην επίμονη ιδέα μια συνεργασία στην παγκόσμια τάξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Έλμαρ Μπρόκ για δύο λεπτά. Δύο λεπτά, δυόμιση λέει ο κύριος Μπρόκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση, αλλά δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσω πάλι νωρίς, διότι στις 10 ε, η ώρα ε, θα συναντηθώ με Τούρκο υψηλό εκπρόσωπο και καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι το θέμα της συνθήκης της Λισαβόνας ε, και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στους διεθνείς οργανισμούς ε, αποτελεί ένα σημείο που υπάρχουν αδυναμίες. Έχει σημειωθεί πρόοδος ε, όταν βλέπουμε την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και το τι ρόλο παίζουν τα ευρωπαϊκά όργανα στα Ηνωμένα Έθνη συντονίζοντας τις θέσεις των κρατών μελών. Είναι σημαντική η δουλειά που γίνεται, αλλά για παράδειγμα όσον αφορά το Ιράν Είδαμε τον ε, ρόλο που έπαιξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή κάποια καλά παραδείγματα, αλλά δεν έχουμε πολύ καλά παραδείγματα σε θέματα όχι θεσμικά αλλά σε θέματα εξουσίας. Αν ε, κοιτάξουμε την ε, ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία και το Ιράκ, τις ε, συνομιλίες της Γενέβης, όταν τελικά φτάσαμε στο θέμα της πάυσης πυρός, οι Ρώσοι προχώρησαν μόνοι τους διότι δεν είχαμε ε, το κύρος που χρειάζεται για να μας πάρουν στα σοβαρά. Αυτό όμως δεν είναι θέμα θεσμικό, αυτό έχει να κάνει με τη δική μας πολιτική και με την ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας μας. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί λόγοι, αλλά νομίζω ότι ο βασικός λόγος είναι ότι στους διεθνείς οργανισμούς ε, έχουμε κάποιες κλασικές διαιρέσεις και ομαδοποιήσεις. Στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τις ανατολικές χώρες. Ε, κάποιες φορές ε, έχουμε προτάσεις από διάφορες ευρωπαϊκές ομαδοποιήσεις, διότι κατά παράδοση υπήρχαν αυτές. Και έχουμε το πρόβλημα ότι τα κράτη-μέλη δεν εγκαταλείπουν τις στρατηγικές αυτές. Ε, έχουμε συνολικά περισσότερα δικαιώματα ψήφου, αλλά καταπολεμούμε ένα τον άλλον. Για παράδειγμα, όταν ε, μιλάμε για τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, των Ηνωμένων Εθνών, βλέπουμε ότι ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας ε, και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήγει σε θέση ώστε τη στιγμή που τουλάχιστον δεν έχουμε μόνιμη θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήγουμε σε μια κοινή απόφαση. Αυτό ισχύει και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μαζί αποτελούμε τη μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να βρίσκεται στην Ευρώπη. Βέβαια, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι υπερβολικό, αλλά στην ε, ε, Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα, εάν πάλι ξεπεράσουμε τις παλιές ε, διακρίσεις και ομαδοποιήσεις, θα γίνει πολύ πιο ισχυρή η θέση μας. Ιδιαίτερα εάν ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε ενωμένοι και ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα. Στο θεσμικό πλαίσιο λοιπόν υπάρχουν ακόμα κάποια ζητήματα όπου πρέπει να γίνουν αλλαγές. Όσον αφορά την πρακτική πολιτική μας έχουμε βελτιωθεί. Είδαμε για παράδειγμα το Ιράν, είδαμε και ε, την ε, διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος ε, στο Παρίσι, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά κατέληξε και συντόνισε την ευρωπαϊκή θέση. Και εάν ξεπεράσουμε τις ε, μεμονωμένες εθνικές μας θέσεις και έχουμε μία κοινή προσέγγιση, θα μας πάρουν στα σοβαρά. Εάν όχι, ε, θα μας ε, χειραγωγούν. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς και έχει να κάνει και με το πλαίσιο και τις ad hoc ή μόνιμες θέσεις στους οργανισμούς αυτούς. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας εδώ και να συζητάμε μεταξύ μας για να καταλήγουμε σε κοινέ δράσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσλέπω στα αποτελέσματα της σημερινής συζήτησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε κατευθείαν στον επόμενο πυρογνώμονα, τον κύριο Ιρμίνσκι. Από ό,τι κατάλαβα θα μιλήσετε για τα εργαλεία, για την ε, ομοφωνία των, σε δράσεις τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών σε διεθνείς οργανισμούς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, ε, έχουμε καθυστερήσει. Αν μπορείτε να είστε σύντομο, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να μιλήσω σύντομα, διότι ήταν πολύ πλήρης η επισκόπηση που ακούσαμε σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξωτερικές πολιτικές και ακούσαμε και για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή φόρουμ. Θα ήθελα εγώ λοιπόν να επικεντρωθώ στα νομικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λοιπόν ε, σύντομα να σας παρουσιάσω κάποιες ε, βασικές ιδέες. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντάς σας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν γιους τρακτάτουμ, δηλαδή αρμοδιότητες στη διεθνή πολιτική δηλαδή την ε, σύναψη διεθνών ε, συνθήκων ε, και τη δυνατότητα να γίνουν μέλη σε διεθνείς οργανισμούς. Ανάλογα βέβαια με το αν ο διεθνής οργανισμός επιτρέπει σε περιφερειακές οργανώσεις όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν μέλη τους. Το πρότυπο για τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών εξαρτάται αφενός από την δομή αυτών των διεθνών οργανισμών, εξαρτάται όμως και από τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά τις εξωτερικές αρμοδιότητες είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος και να συμμετέχει σε, αυτές, σε αυτούς τους οργανισμούς εφόσον επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μέλος. Μόνο δηλαδή σε περίπτωση που λένε ότι μόνο τα κράτη-μέλη ε, μπορεί να είναι μέλη, ε, δεν μπορεί να συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τι ε, κοινέ αρμοδιότητε, τι μοιρασμένε αρμοδιότητε, εδώ είναι διαφορετική η κατάσταση. Τα κράτη-μέλη είναι τα βασικά συμβαλόμενη μέρη και κατόπιν ε, είτε συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή αντικατέστησε ε, τα κράτη-μέλη στις εξωτερικές πολιτικές. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ ε, στις Στι ε, ρήτρε ε, σχετικά με τη δευτερεύουσα θέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικά μοντέλα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πρώτη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδρυτικό μέλος ή στη δεύτερη περίπτωση προσχωρεί αργότερα, μετά δηλαδή τα κράτη-μέλη τη. Συχνά επίσης έχουμε κοινέ συμφωνίε, δηλαδή Έχουμε συμφωνίες ε, που έχουν να κάνουν με τις ε, μοιρασμένες εξωτερικές αρμοδιότητες. Ε, χρήσιμο για τις περαιτέρω συζητήσεις είναι η ιδέα ότι οι διεθνείς συμφωνίες συνάπτονται στο όνομα των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δηλαδή προηγούμενη συμμετοχή των κρατών μελών και οι αρμοδιότητες τους ε, κατόπιν ε, έχουν γίνει αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λόγω των εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική. Όσον αφορά το δικαίωμα ψήφου που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παρουσίαση του κυρίου Βότερ, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα να έχουμε ξεχωριστά δικαιώματα ψήφου, αλλά με κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε κοινό δικαίωμα ψήφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει δηλαδή στο όνομα των κρατών μελών. Το άλλο πρότυπο για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι διεθνείς συμφωνίες ε, που ε, συνάπτονται υπό την αιγίδα ε, μιας διακυβερνητικής οργάνωσης ή έχουμε μικτές περιπτώσεις. Το ένα παράδειγμα ήταν αυτό που μόλις ανέφερε ο κύριος Μπρόκ, η Συμφωνία του Παρισιού το 2015 στο πλαίσιο της σύμβασης πλαίσιο της, των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που υιοθετήθηκε μετά την διάσκεψη των μερών στο Παρίσι. Εδώ λοιπόν ε, έχουμε μια μεικτή κατάσταση, διότι είχαμε την ε, μεικτή απόφαση στην διάσκεψη των μερών και κατόπιν είχαμε την συμφωνία, η οποία είναι μια ξεχωριστή διεθνή συμφωνία, η οποία πρέπει πρώτα να υπογραφεί και να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με του τους ε, εσωτερικούς κανόνες της συνθήκης δηλαδή όσον αφορά ε, τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις ε, των ε, διεθνών διακυβερνητικών οργανώσεων όπως ανέφερα, έχουμε δύο ξεχωριστά πρότυπα. Έχουμε συντονισμένες πολιτικές και μη συντονισμένες πολιτικές, ε, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασκεί τα δικαιώματα των κρατών μελών. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη για συντονισμός με την νομική έννοια, υπάρχει μόνο ανάγκη για ομοφωνία ε, και συμμόρφωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν έχουμε τα κοινά δικαιώματα ψήφου, ε, που δεν είναι επίσημος νομικός όρος. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε δικαιώματα ψήφου των κρατών μελών εντός των ε, διεθνών οργανισμών ε, που ασκούνται όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα των κρατών μελών. Και αυτό συμβαίνει συχνά όταν έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αρμοδιότητας που έγινε αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δευτερεύουσες νομικές πράξεις ε, που καθιστούν απαραίτητη την κοινή δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν έχουμε ξεχωριστή ψήφο, ε, έχουμε τις, ε, κοινές, τις μικτές συγγνώμη, συμφωνίες. Επίσης είναι δυνατός ο συντονισμός πολιτικών εντός των διακυβερνητικών οργανισμών και σε περίπτωση αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας των κρατών μελών. Υπάρχει η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να απέχουν από την ψηφοφορία. Αυτό συμβαίνει όταν δεν συμπεριλαμβάνεται ρήτρα για την κοινή ψήφο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ψηφίζουν ομόφωνα σε περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συμμετέχει αλλά δεν έχει δικαίωμα να ασκεί το δικαίωμα ψήφου των κρατών μελών. Και, καταλήγω το, και φτάνω τώρα στο κεντρικό ε, μέρος της παρουσίασής μου. Έχει να κάνει με την ψήφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα των κρατών μελών. Ε, διάφοροι διακυβερνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάπως ιδιαίτερη περίπτωση διότι μπορεί να αναφέρεται ως η μόνη περιφερειακή οργάνωση που αποτελεί συμβαλόμενο μέρος σε μιας ε, συνθήκης. Ε, Είναι απαραίτητο λοιπόν να διασφαλιστεί η συντονισμένη δράση. Ένα παράδειγμα είναι ε, το άρθρο 9 της ε, συμφωνίας ε, που καθιερώνει τον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Τότε βέβαια είχαμε ευρωπαϊκές κοινότητες ε, αντί για Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν όμως το δικαίωμα να ασκούν το δικαίωμα ψήφου των κρατών μελών ε, που από τη μεριά τους θα έπρεπε να απόσχουν. Τώρα λοιπόν έχουμε 28 ψήφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί για 28 ψήφους των κρατών μελών που θα μπορούσαν να διαφέρουν μεταξύ τους. Όπως ε, ήδη αναφέρθηκε, υπάρχει το πρόβλημα οικοδόμησης περιφερειακών συνασπισμών Ε, λόγω της ε, μειοψηφίας που αντιπροσωπεύουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αλλά ήθελα να σας δώσω το παράδειγμα αυτό. Υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα, ιδιαίτερα στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Για παράδειγμα, η ρήτρα στην Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Σημαντικό είναι επίσης ε, και είναι καθαρά νομικό το θέμα αυτό. Κάποιε από τις ρήτρε επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ασκούν τα δικαιώματά τους. Και στην περίπτωση αυτή ο Περιφερειακός Οργανισμός δεν μπορεί να ασκεί το δικαίωμα στο όνομα ε, του κράτου μέλου ή άλλων κρατών μελών. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ένα κράτο μέλο θέλει να ενεργήσει ξεχωριστά, χωρί συντονισμό των δράσεων. Αυτό ε, δεν εκτιμάται, ιδιαίτερα λαμβάνοντα υπόψη το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Ε, ενδιαφέρουσα λοιπόν είναι η δυνατότητα να επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα στο όνομα των υπολείπων κρατών μελών. Επίση, σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι σε κάποιες ε, περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να ε, ψηφίσει ανάλογα με τον αριθμό των κρατών μελών που είναι συμβαλόμενα μέρη. Ένα παράδειγμα είναι η Σύμβαση του Ελσίνκη για την ε, προστασία του περιβάλλοντος στην ε, Βαλτική. Επίση, είναι δυνατόν να περιοριστούν οι ψήφοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράδειγμα εδώ είναι η ΚΟΤΙΦ η Διεθνή Συμφωνία για τις Μετακινήσει. Μετακινήσεις. Ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες ε, στον τομέα των μεταφορών. Από τη μία μεριά υπάρχει δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ψηφίζει στο όνομα των κρατών μελών, ενώ σε άλλους τομείς πρέπει τα κράτη-μέλη να ψηφίζουν. Ένα παράδειγμα των προβλημάτων που μπορεί να έχει κανείς. Όταν έχουμε την ε, μεικτή διαδικασία μιας απόφασης ε, και σύμβασης. Ε, έχουμε την Συμφωνία του Παρισιού από την διάσκεψη των μερών στο Παρίσι. Γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας διεθνής οργανισμός και υπάρχει εδώ μια διεθνή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Ανέφερε το παράδειγμα αυτό και ο κύριος Πρόκ. Ένα από τα κράτη ήταν η Πολωνία που υπέβαλε δήλωση σχετικά με την, ε, την συμμετοχή του σύμφωνα με το πρωτοκόλλο του Κιώτο. Είναι σημαντικό όμως να γνωρίζουμε ότι αν έχουμε ξεχωριστή συμφωνία που υιοθετείται από ένα διεθνή οργανισμό ή από την ε, διάσκεψη των μερών, τη EOP, τότε ξεκινούν τα προβλήματα όταν έχουμε δηλαδή μια διεθνή συμφωνία η οποία θα πρέπει να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη. Εναλλακτική μέθοδος ε, είναι η έννοια των subordination clauses είναι ρήτρε που συμπεριλαμβάνονται στις διεθνείς ε, συμφωνίες που επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλους διεθνού οργανισμούς, αλλά στην πράξη μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να, ε, ε, την, να υπογράφουν τη συνθήκη μόνο μετά από προσχώρηση όλων ή συγκεκριμένου αριθμού των κρατών μελών της. Αυτό είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί τα κράτη αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, βοηθάει τη... τους διεθνείς οργανισμούς περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έβρισκε τρόπο αλλά είναι τρόπος ώστε να έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μέλος μόνο εφόσον όλα ή συγκεκριμένο αριθμός των κρατών μελών προσχωρεί. Και στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη θέση των κρατών μελών, δεν θα υπάρχουν μεμονωμένες θέσει των κρατών μελών. Αυτή η ρήτρα λοιπόν συνοδεύεται και από την κοινή, τη ρήτρα για την κοινή ψήφο διότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στον διεθνή οργανισμό, είναι δυνατόν να ασκεί το δικαίωμα ψήφου των κρατών μελών. Προφανώς δεν υπάρχει κάποιος ε, κανόνας που να ρυθμίζει αυτήν ε, την ρήτρα είναι όμως χρήσιμος μηχανισμός ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργεί σε συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Όλες οι δευτερεύουσες πράξεις θα πρέπει να συνάδουν με το διεθνές δίκαιο, που είναι το δίκαιο που απορρέει από αυτόν τον διεθνή οργανισμό. Και επειδή τα κράτη-μέλη είναι και αυτά μέλη του διεθνούς οργανισμού, δεν ε, θα υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε αυτές τις δύο νομικές ρυθμίσεις. Ο όρος subordination clause, ρήτρα υποταγής, περιέχει τη λέξη υποταγή, αλλά δεν υποτάσσεται κανείς σε κάποιον άλλον. Ε, απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποχρεώνεται να εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Αυτά μπορώ να σας τα δείξω με κάποια παραδείγματα, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχουν ε, πολλοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο, για παράδειγμα οι περιφερειακοί οργανισμοί διαχείρισης αλληλείας, όπου συμμετέχουν τα κράτη-μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούν τα κράτη-μέλη να υποβάλουν δήλωση για την εδαφική εφαρμογή. Έχουμε για παράδειγμα το άρθρο 13 της σύμβασης ICAT που λέει ότι όταν ένας οργανισμός ε, γίνεται συμβαλόμενο μέρος της σύμβασης αυτής, τα κράτη-μέλη του οργανισμού αυτού πάβουν ε, να είναι συμβαλόμενα μέρη της σύμβασης θα γίνεται γραπτή κοινοποίηση στον ε, Γενικό Γραμματέα του ΦΑΟ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι απαραίτητο να εγκαταλείψουν ε, την ε, θέση τους τα κράτη-μέλη στον Διεθνή Οργανισμό και να παραχωρήσουν τη θέση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά παραδείγματα είναι η UNCLOS, η Σύμβαση για τη Θάλασσα και πάλι σας αναφέρω το παράδειγμα της Σύμβασης COTIF. Υπάρχουν ε, επίσης προβλήματα με τις ε, ρήτρες υποταγής αυτές. Ένα από τα ζητήματα που τίθενται είναι αν είναι απαραίτητη ε, μια ρήτρα υποταγής για να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν τον ε, συγκεκριμένο διεθνή οργανισμό. δεν είναι απαραίτητο και πολύ συχνά συμπεριλαμβάνονται αυτές οι διεθνείς ε, συμφωνίες στις συνθήκες προσχώρησης. Έτσι ρυθμίζεται η αρμοδιότητα. Και η δική μου θέση είναι ότι οι ρήτρε υποταγή μπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικό τρόπο εφαρμογή του άρθρου 351 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέει ότι οι διεθνεί υποχρεώσει των κρατών μελών συνεχίζουν να ισχύουν μετά την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η δεύτερη παράγραφο ε, αναφέρει ρητά ότι τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με την νομική τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι συνήθως πρέπει να, ε, ε, να αποχωρούν από τις ε, συνθήκες. Κλείνοντας λοιπόν να πω ότι πρέπει να ε, εξετάσουμε την ε, διαδικασία για τη σύναψη διεθνών ε, συμφωνιών από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των κρατών μελών να ελέγχουν τη διαδικασία αυτή. Όπως σας είπα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών. Ένα από τα παραδείγματα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, των Ηνωμένων Εθνών. Το άλλο είναι ο Διεθνής Οργανισμός ε, Εργασίας, όπου έχουμε συμμετοχή αποκλειστικά των κρατών μελών. Σημαντικό είναι να τονιστούν οι μηχανισμοί της συνθήκης που προβλέπουν ε, συμμόρφωση και άλλωστε υπάρχει και το θέμα του μη υποχρεωτικού δικαίου που έχει να κάνει με την με τις κοινέ πολιτικές εντός των διακυβερνητικών οργανισμών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μοιρασμένων αρμοδιοτήτων. Αυτά για τώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η Πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και τώρα ευθύ αμέσω να δώσουμε το λόγο τον κύριο Γιώνα Τζόνσον, ο οποίο είναι τμήματάρχη στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για τι Πολυμερεί Σχέσει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα προσπαθήσω να εξετάσω το θέμα της ε, πρακτικής εφαρμογής του, του θέματος τους ε, πολυμερούς εκπροσώπησης. Ο κύριος ε, Βάουτερς ανέφερε την υπάτη εκπρόσωπο κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη η οποία απευθύνθηκε προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επρόκειτο για κάποια ομιλία της που ήταν πολύ περιεκτική και ενδιαφέρουσα συζήτηση που επικολούθησε ε, και έχω να σας ε, συστήσω αν μπορέσετε να διαβάσετε αυτήν την ε, ομιλία της κυρίας Μογκερίνη διότι φάνηκε με συγκεκριμένο τρόπο το πώς συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο έργο των Ηνωμένων Εθνών για τα διάφορα προβλήματα του κόσμου αναφέρθηκε η Συρία, είμαστε ο πρώτος ε, δωρετής, αναφέρθηκε η Λιβύη. Και ε, απόψε εγκρίθηκε το ψήφισμα 2292 για την επιχείρηση ε, Σόφια που αφορά την Λιβύη και το ε, την, την ε, ασφάλεια κατά θάλασσα. Είναι την ο πλευρό ασφαλεία, πολύ σημαντικό το απόψινο ψήφισμα. Τώρα, όσον αφορά ε, άλλε διασκέψει που ανέφερε, ήταν η διάσκεψη για το Αφγανιστάν του Οκτωβρίου και επίσης την εταιρική σχέση για το μεταναστευτικό που και αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι φαίνεται το ότι σήμερα περισσότερο παρά ποτέ χρειάζεται ε, πολυμερής διπλωματία. Χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ. Και βλέπουμε ότι συνεχώς ε, ενλύνεται η συνεργασία με τον ΟΗΕ. Αναφέρθηκε για το COP21 το 2015 πάντως, έχουμε και άλλες σημαντικές εξελίξεις, αλλά και συμφωνίες πρώτα-πρώτα, το θεματολόγιο του 2020 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεύτερον, τις αξιολογήσεις για την ειρήνευση, για τον ρόλο της γυναίκας και το ψήφισμα 2025 και όσον αφορά το θεματολόγιο του 2030 χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποσπάστηκε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για την ε, χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου σε σχέση με ε, την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να υπάρξει αξιολόγηση ε, ειρήνευσης και προστασίας στο αμάχου πληθυσμού δεν πετύχαμε όλα όσα θέλαμε, αλλά ήταν σημαντική συμβολή ε, στη συζήτηση και σε αυτές τις αξιολογήσεις και αναθεωρήσεις και για το COP21 που αναφέραμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και το αποτελέσμα ήταν πολύ θετικό. Όλα αυτά θα έχουν σημασία ε, για το μέλλον και θα πρέπει τώρα να δούμε τι υλοποιήστε για αυτών των συμφωνιών. Γι' αυτό το 2016 είναι σημαντικό έτος. Και τον Ιούλιο το Συμβούλιο θα αποφασίσει το ακριβώς τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να ελοπίσει τα συμφωνηθέντα. Επίσης, αυτές οι μεταρρυθμίσεις πολύ σημαντικές για τη σχέση μας με τον ΟΗΕ. Αυτά τα θετικά αποτελέσματα τα πετύχαμε γιατί η φωνή μας ήταν ενιαία. Ξέρουμε ποιε είναι οι προκλήσει, ποια είναι τα προβλήματα όσον αφορά την εξωτερική εκπροσώπηση. Αλλά θα πρέπει να τονίζουμε και τα θετικά, όχι μόνο τι δυσκολίε. Η συνθήκη τη Λισαβόνα είναι μια πολύ χρήσιμη αφετηρία και βάση. Αυτά όπως τονίστηκαν ε, οδήγησαν στην ε, αναβάθμιση του, των δικαιωμάτων της εκπροσώπησης και συμμετοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ε, ΟΗΕ για την ΆΝΚΑ όπου μπορέσαμε πάλι να αναβαθμίσουμε τον ρόλο μας και την 6η Ιουνίου ε, συμμετείχαμε στις συζητήσεις περισσότερο από ό,τι πριν. Και όπως αναφέρθηκε, σε καθημερινή βάση υπάρχει συντονισμός. Στην Νέα Υόρκη, στις ε, αντιπροσωπίες Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται και χίλιες συναντήσεις ε, ετησίω ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ενιαία φωνή για όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ σε 90% ε, των περιπτώσεων πετυχαίνουμε κοινή τοποθέτηση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και τα κρατημέλη βέβαια που έχουν κάποιο ρόλο, δεν είναι μόνο η αντιπροσωπεία. Ε, και τα κρατημέλη ακριβώς, έχουν συμφέρον προς τούτο και συγκριτικό πλεονέκτημα στις Βρυξέλλες επίσης με διαφορετικές ε, μεθόδους ε, γίνονται προπασκευαστικές κινήσεις όπως για το θέμα του 2030 και στο Συμβούλιο επίσης υπάρχουν κάποιες ομάδες εργασίας ε, προετοιμάζουν τις διεθνείς επαφές μας και την προσαρμογή μας στις διαπραγματεύσεις. Οι συντονιστικές προσπάθειες ακριβώς όπως ελέγχθη είναι δύσκολες και θα πρέπει να εντείνουμε τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες αλλά αποδείχθηκε από τις για την Agenda 2030 ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Επομένως φάνηκε το τι μπορούμε να πετύχουμε όπως και σε Παρίσι, Γενέβη, Ναϊρόμπι, Ρώμη όλες μας οι αντιπροσωπείες ε, έχουν πάρα πολύ θετικό ρόλο και έτσι συντονίζονται οι θέσεις των κρατών μελών ε, για τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν έδρα στις πρωτεύουσες που σας προανέφερα. Οι προσπάθειες δεν σταματούν για να βελτιωθεί το στάτους μας στους διεθνείς θεσμικούς οργανισμούς. Πολλές φορές υπάρχει κάποιο εσωτερικό φρένο σε σχέση με το μέχρι που θα φτάσουμε όσον αφορά την υιοθέτηση κοινή θέση για τις κοινέ αρμοδιότητες και από την άλλη μεριά ε, έχουμε τις αρμοδιότητες του κάθε κράτους μέλους. Εδώ πηξίδα μα είναι η συνθήκη, αλλά πολλές φορές χρειάζεται να γίνουν και σχετικές ζυμώσει και συζητήσει. Επίση, κάποιε τρίτε χώρε είναι καλοί μας σύμμαχοι, φίλοι και έχουν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τοποθετείται, να εμφανίζεται σαν μπλοκ ενιαία. Ε, τα, αναφέραμε τα σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου. Ε, λέμε ότι είμαστε ενιαίο μέτωπο, θα έχουμε μία ψήφο ή 28 ψήφους όσο και τα κράτη-μέλη αυτή η προβληματική υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, οι ίδιοι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον θα αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας τους και αν ακριβώς ε, συμμορφωθούν, να συντονιστούν με τόσα ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα υπάρχουν παρόμοια αιτήματα από παντού. Γι' αυτό πολλές φορές τα πράγματα γίνονται διακριτικά. Ε, υπάρχει ιδιαίτερη μεθοδολογία. Σε κάθε διεθνή οργανισμό που προσπαθούμε τα δικαιώματα συμμετοχής μας να τα αναβαθμίσουμε. Δεν ξεχνούμε ποια είναι τα προβλήματα, και το θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ρεαλιστικά. Πάντως, για να επανέλθουμε στα θέματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα πρέπει να έχουμε ενιαία τοποθέτηση. Ιδίως εκεί, στον ΟΗΕ. Και τα πλευρά προβλήματα θέλουν πολυμερή αντιμετώπιση. Είμαστε από τους πιο ε, καλά οργανωμένους διεθνούς φορείς και ούτως ώστε μπορούμε να κάνουμε τη φωνή μας να ακούσει στον ΟΗΕ. Αλλά ταυτόχρονα βοηθούμε και τον ΟΗΕ. Τον βοηθούμε να βελτιώσει τις επιδόσεις του στην διεθνή σκηνή. Και εμεί επομένω προσπαθούμε συνέχεια να βελτιωθούμε όσον αφορά την αποτελεσματικότητά μα ε, στα πλαίσια της ε, διεθνού τάξης και σκηνή. Η πρόεδρο, ευχαριστώ. 15 λεπτά μας μένουν για την συζήτηση. Πρώτα ο Χαμών Χαουρέγγι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα πρώτα πρώτα να ορίστε να σας μιλήσω στα ισπανικά, ε, φορές τα ακουστικά σας. Ξαναρχίζει ο Γιώργος Χάουρικη. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτό το οποίο είπατε. Πρόκειται για μια προβληματική που ανάγεται στο παρελθόν και κρατάει χρόνια. Η κυρία Μογκερίνη νομίζω ότι έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στην ε, εξέλιξη της διεθνούς πολιτικής και εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Εκεί επίσης θέλω να σας επισημάνω το εξής. Πεςτε μου τη γνώμη σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, ξέρετε, πολλά εσωτερικά ζητήματα απαιτούν πιο δυναμική εξωτερική πολιτική. Θέλω να πω το ότι έχουμε τώρα κάποιους στόχους πολύ σημαντικούς για την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε μια ισχυρή εξωτερική πολιτική για να σας πω κάποια παραδείγματα που θα σας δείξουν τι εννοώ πρώτα πρώτα το προσφυγικό και η σχετική πολιτική μας εγώ νομίζω ότι η Ευρώπη για να δώσει μια λύση στο προσφυγικό και στη σχετική κρίση αυτό θα γίνει μόνο εάν υπάρχει μια εξωτερική και διεθνής πολιτική που θα εξασφαλίζει την διεθνή αλληλεγγύη. Βέβαια δεν έχουμε καν αλληλεγγύη στο εσωτερικό της Ένωσης. Και οι διαστάσεις του προσφυγικού είναι τέτοιες που ξεπερνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε απαιτούνται αποφάσεις σε εθνές επίπεδο. Γι' αυτό και εγώ σας λέω ότι χρειάζεται μια Ευρωπαϊκή Ένωση με πυγμή σε εθνές επίπεδο, με πυγμή ε, στα πλαίσια και στο, στην πλατφόρμα του ΟΗΕ, ούτω ώστε να βρεθούν οι λύσεις στα δικά μας εσωτερικά προβλήματα. Άλλο ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτό το καμπανάκι κινδύνου που έχει χτυπήσει για την φοροδιαφυγή. Εδώ και ένα χρόνο ε, συζητάμε έντονα το πρόβλημα. Έχουμε δύο εξεταστικές επιτροπές, την TAX 1 και TAX 2 και από το Σεπτέμβριο θα συγκροτήσουμε και μια ερευνητική επιτροπή για τα Panama Papers. Θα κρατήσει αυτή η θητεία αυτών των επιτροπών ένα χρόνο. Οπότε για τους εταιρικούς φόρους ε, για την καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής μέσω των φορολογικών παραδείσων. Όλα αυτά ε, απαιτούν συνεργασία σε διεθνές επίπεδο. Στον ΟΣΑ και στο δόνο του. Επομένως, μόνο έτσι θα βρούμε κάποιες λύσεις. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι για να λύσει τα δικά της προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει πιο δυναμικό διεθνές ρόλο. Τρίτο και τελευταίο, θέλω να σας πω κάτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνοηθεί και συντονιστεί περισσότερο με την υπάτη εκπρόσωπο. Μια που κάθε, σε κάθε ολομέλεια ε, αναλύουμε τρεις ε, βασικές χώρες, τρεις βασικούς τόπους με προβλήματα ε, από όλο τον κόσμο. Και αυτό γίνεται και στις κοινοβουλικές επιτροπές. Δηλαδή, ε, είμαστε σαν, σαν ένας ε, φάρος, φωτοδότης για όλο τον κόσμο, για αυτό το μέτωπο. Οπότε θέλουμε να υπάρχει κάποιο είδους σύνδεση αυτών των προσπαθειών με τις προσπάθειες διεθνούς εξωτερικής πολιτικής μας, ιδίως στον ΟΗΕ και άρα το θέμα δεν είναι το να τονίζουμε, το να διεκδικούμε τις μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το πώς η νέα φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακούγεται πιο ισχυρή σε προβλήματα, προβλήματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης και της παγκοσμιοποίησης. Και γι' αυτό σας λέω ότι τα όσα μας συστήσατε ε, βοηθούν προς όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα και θα ήθελα εγώ να πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτά. Και εγώ θέλω να, λέει λέει ίδια η πρόεδρος, να κάνω ένα σχόλιο και να κάνω μια ερώτηση. Θα έχετε ακούσει ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω εδώ στην Επιτροπή Συνταγματικών επεξεργαζόμαστε μια πρόταση για καλύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ε, νέα συνθήκη για θέματα ε, κοινή εξωτερική πολιτική κτλ. Οι αδυναμίε στι οποίε αναφερθήκατε και εσά, οι αδυναμίε λειτουργία μα, Εκεί χωρεί ακόμα βελτίωση και στην βάση της υφιστάμενης συνθήκης, η οποία συνθήκη ούτως ή άλλως βελτίωσε το καθεστώς και της παρουσίας της Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Είμαστε ενισχυμένοι παρατηρητές τώρα. Νομίζω ότι καλά τα πάμε στο, στη Νέα Υόρκη, λιγότερο καλά στον FAO για παράδειγμα στον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων. Ερώτηση λοιπόν, βλέπετε δυνατότητα βελτιώσεως στον συντονισμό ή και σε, άλλες, σε άλλους τομείς λειτουργίας μέσα στα πλαίσια της παρούσας συνθήκης και για τη συμμετοχή μας σε διάφορους άλλους διεθνείς οργανισμούς και στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποια στιγμή θα αναθεωρηθεί η συνθήκη. Εάν αναθεωρηθεί η συνθήκη ποιες θεωρείτε ότι θα ήταν οι τομείς, ποιοι θεωρείτε ότι θα ήταν οι που θα έπρεπε να ρίξουμε ιδιαίτερο βάρο, για παράδειγμα συμμετοχή στο Συμβούλιο ασφαλεία, Πού βλέπετε ότι θα έπρεπε να γίνουν κάποιε θεμελιώδει αλλαγέ, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολυμερή πλαίσια και βέβαια υπό την ισχύ του παρόντο καταστατικού χάρτου των Ηνωμένων Εθνών. Πού θεωρείτε λοιπόν ότι θα μπορούσαν να γίνουν αλλαγέ, αλλά και εκεί γιατί <clears throat> ακόμα στην ουσία λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο των εποχών του ψυχρού πολέμου. Αυτή είναι η μία ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Ακούγοντας τον πρέσβη μας στα Ηνωμένα Έθνη και ακούγοντας εσάς, δεν είναι σαφές για μένα τι και πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας μέσα σε διεθνείς οργανισμούς διά της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Πόσα μπορούν να γίνουν μέσω των δομών που έχουμε στην ε, διπλωματική μας αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη Μπορεί να βελτιωθεί ο συντονισμός. Υπάρχουν άλλα αμφιλεγόμενα ζητήματα ή διαχωριστικές γραμμές και είπατε και μια φορά ότι λόγω έλλειψης δυνατότητας συντονισμού αλλά και λόγω της διστακτικότητας των χωρών μελών να αυτοϋπαχθούν σε κάποιες προσπάθειες συντονισμού γιατί προτιμούν να μιλούν για λογαριασμό τους. Πώς ενισχύεται η δύναμή μας όταν λέτε ότι άλλες χώρες όπως κάποιες γειτονικές μας χώρες αλλά και η Νορβηγία για παράδειγμα συμπαρατάσσονται μαζί μας. Αυτό έχει κάποια ορατή απήχηση στην αύξηση της δύναμης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για πρόβλημα ή πρόκειται για ε, ένα πλεονέκτημα. Γιατί είπατε κύριε και καμιά φορά πώς μας βλέπουν άλλες χώρες. Αν μπορείτε λοιπόν παρακαλώ να σχολιάσετε τα θέματα αυτά. Άλλος κανείς από εκ των συναδέλφων. Όπως θέλετε να απαντήσετε, με όποια σειρά θέλετε. Εφτά λεπτά μας μένουν. Ο κύριος Βάουτερς, καθηγητής. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες και σημαντικές ερωτήσεις σας. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι αρχικές μας αντιδράσεις είναι αντιδράσεις επιτόπου. Ίσως να χρειαστεί κάποιος χρόνος προβληματισμού για να αντισκεφτούμε καλύτερα τις ερωτήσεις αυτές. Στην Ευρώπη μας αρέσει να αλλάζουμε τις συνθήκες μας. Αυτό είναι μέγα πλεονέκτημα και είναι και η μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Όμως, στην σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση με τις 28 χώρες μέλη, το έδειξε και η διαδικασία κύρωσης της ε, Συνθήκης Λισαβόνας, είναι δύσκολο να αναθεωρηθούν. Άρα, πρώτη απάντησή μου. Ας βελτιώσουμε τη λειτουργία της υφιστάμενης συνθήκης. Ήδη έχουμε έξι χρόνια που λειτουργούμε υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορεί να γίνει κάποια πιο συστηματική καταγραφή των ε, επιτευμάτων και στα Ηνωμένα Εθνή και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς. Να μην δυσμονούμε ότι υπάρχει πραγματικότητα των συνθήκων, υπάρχει πραγματικότητα της πρακτικής μας επιτόπου, εντός δηλαδή των διεθνών αυτών οργανισμών, αλλά υπάρχουν και οι ταχύτατες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον ο κόσμος ε, δεν παραμένει ακίνητος. Σημειώθηκαν τόσες κρίσεις. Αναδύονται άλλες δυνάμεις και μάλιστα με όλο και δυνατότερη φωνή και που ε, ζητούν να έχουν περισσότερα δικαιώματα συμμετοχής οι ίδιες σε διεθνείς οργανισμούς εξακολουθούν να επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έχουν κάπου και δίκιο ότι παρά είναι πολλοί Ευρωπαίοι στις αίθουσε των διεθνών οργανισμών. Δεν δέχονται την ιδέα ότι θα πρέπει να αναβαθμίζεται διαρκώς η θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς να υπάρχει από την άλλη μεριά μια προσαρμογή της θέσης των χωρών μελών. Αυτό είναι ευαίσθητο θέμα, το οποίο μάλιστα έχει οδηγήσει και σε δύσκολες διαπραγματεύσεις στην Γενική Συνέλευση. Θα πρέπει διαρκώς να ζητούμε περισσότερα ή θα πρέπει κάπου και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει κάποιες ευθύνες. Νομίζω ότι μέσα στην παρούσα πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει. Όμως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τρίτε χώρε σε ό,τι αφορά την θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνεί οργανισμού. Και χωρί να λησμονούμε ότι οι διεθνεί οργανισμοί του οποίου συζητούμε εδώ έχουν παραχθεί όλοι από δικέ μα προσπάθειε. Και τώρα αυτέ οι αναδυόμενε δυνάμει προσπαθούν να αλλάξουν του οργανισμού αυτού από μέσα. Και αν δεν το επιτυγχάνουν αυτό, βλέπουμε χώρε όπω η Κίνα να, που πηγαίνουν και φτιάχνουν νέους διεθνείς φορείς, όπως η Κινέα για παράδειγμα που φτιάχνει την ε, Παγκόσμια Ασιατική Τράπεζα. Ε, το ζήτημα είναι πώς θα ανταποκριθούμε εμείς σε αυτό, πώς θα απαντήσουμε εμείς. Δυστυχώς, οφείλω να ομολογήσω ότι σε αυτή την Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα εμείς ανταποκριθήκαμε με πραγματικά πολύ λάθος τρόπο. Αποφάσισαν 15-16 χώρες να πάνε να συμπαραταχθούν με αυτή την τράπεζα χωρίς να υπάρχει συντονισμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να συνεργαστούμε όχι μόνο με τα Ηνωμένα Έθνη, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε και μια στρατηγική απάντηση δική μας. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει στρατηγικό σχεδιασμός και να συνταχθεί και στρατηγικό έγγραφο για το πώς επιθυμεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους διεθνείς οργανισμούς. Θα θυμίστε ότι το 2012 εξεδόθη ανακοίνωση από, από τον τότε πρόεδρο της Κομισιόν Βαρόσο στην οποία η Λέδη Άστον, ως είπατε εκπρόσωπος τότε, έκανε ένα είδους στρατηγικό εγχείρημα. Δηλαδή, ποιους διεθνείς οργανισμούς θέλουμε, σε ποιους οργανισμούς θέλουμε να ενισχυθεί ή να αναβαθμιστεί η θέσεις μας. Δεν συζητείται πλέον αυτό το έγγραφο, δεν γνωρίζουμε τι κάνει ακριβώς με το θέμα αυτό η Επιτροπή Juncker αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει ένα σχέδιο να μπουν προτεραιότητες και ένα χρονοδιάγραμμα δηλαδή τι θέλετε να επιτύχετε και πότε ή έως πότε κάτι που είναι επίσης σημαντικό είναι να γίνει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σχεδιασμό της στρατηγικής της αναβάθμισης της θέσεως της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, στους διεθνείς οργανισμούς. Είναι δύσκολο το περιβάλλον και εσωτερικά και εξωτερικά. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική θα συνεχίσουμε να κινούμαστε ασυντόνιστα και αυτό πάντως όχι προς όφελός μας. Αυτή είναι η θέση μου για τα πράγματα αυτά και πολύ ευχαρίστω να επεκταθώ εφόσον το επιθυμείτε. Yes, thanks. Ευχαριστώ. Καταρχάς, στον Ευρωβουλευτή που πήρε το λόγο, να πω ότι συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να φροντίσουμε το θέμα της μετανάστευσης, που τέθηκε ως παράδειγμα, να έχει υψηλή θέση στο θεματολόγιο του ΟΗΕ. Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι παγκόσμιο. Δεν αποτελεί πρόκληση αποκλειστικά για την Ευρώπη και θα είναι καλή ευκαιρία να το θέσουμε στην ε, διάσκεψη κορυφής για τη μετανάστευση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο. Το θεματολόγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως ε, είπα, αποτελεί σημαντικό επίτευγμα. Έχουμε και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που αποτελούν σημαντική επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θεματολόγιο παγκόσμιας διακυβέρνησης, διεθνούς διακυβέρνησης ε, και είναι κάτι που συμπεριλαμβάνει όλες ε, τις ε, παγκόσμιες προκλήσεις συμπεριλαμβανομένης τη μετανάστευση. Νομίζω ότι πάντα αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησή μας. Ποιε είναι οι πολιτικέ μας, τι θέλουμε να πετύχουμε και πόση επιτυχία έχουμε στην επίτευξη των στόχων αυτών. Έχουμε τη συνθήκη μας, θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε, θα πρέπει να την αναπτύξουμε προφανώς, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει και εσωτερικά να πείσουμε όχι μόνο Πρέπει να πείσουμε τους ε, ενδιαφερομένους κύκλους ε, στις χώρες μας ότι η προστιθέμενη αξία αυτή είναι προστιθέμενη αξία και για τις χώρες μας και σε τομείς ε, της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας μπορούμε να δείξουμε ότι θα έχουμε περισσότερο αντίκτυπο ενωμένοι και θα μπορέσουμε να πείσουμε όλους τους ενδιαφερομένους όπως νιώθω ότι κάναμε στις διαπραγματεύσεις μας για την Ατζέντα 2030 όπου είχαμε πολλή υποστήριξη από τα κράτη-μέλη μας. Πρέπει να δείξουμε πώς σε, ευρωπαϊκ... πώς σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε να επιφέρουμε τη θέμενη αξία. Θα πρέπει να σχηματίσουμε διεθνείς συνασπισμούς ώστε να συνεργαστούν μαζί μας και άλλες χώρες στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. δεν θέλουμε απαραίτητα δημιουργία νέων οργανισμών, ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το διεθνές πλαίσιο που υπάρχει. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση όσον αφορά την τυπική μας θέση στους διεθνείς οργανισμούς ε, και τα δικαιώματα συμμετοχής μας. περιέγραψα κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε εξετάζοντας κάθε περίπτωση ανάλογα με τον οργανισμό, ανάλογα με την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται, για να δούμε πώς μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Φυσικά θα χαρούμε να συνεργαστούμε με όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβάνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για να δούμε πώς μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους του Έλμαρ Μπρόκ που έπρεπε να αποχωρήσει. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση αυτή. Μπορούμε τώρα να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις δυνατότητες της ε, υπάρχουσας ε, συνθήκης της σα συνθήκη. Και επίση ε, βελτιώνουμε τη δυνατότητα αντίδρασής μας ε, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σημαντικό είναι να είμαστε αποτελεσματικοί στο διεθνές πλαίσιο και Ζητώ συγγνώμη, άρχισα να συνοψίζω χωρίς να σας δώσω το λόγο. Ζητώ συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα απλά να πω λίγα λόγια. διότι αναφέρατε τις χώρες που επιθυμούν στενότερη συνεργασία με την Ρωσία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι σημαντικό για την Ένωση να καθορίσει τους στόχους της στην διεθνή πολιτική. Χρειαζόμαστε κάτι σαν οδικό χάρτη σχετικά με το πώς θα εφαρμόσουμε την πολιτική αυτή και στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε την ε, ενισχυμένη συνεργασία. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη διπλωματία μας για να ενισχύσουμε τη θέση μας και να καταστήσουμε σαφείς τις θέσεις μας. Ε, θα υπάρχουν όμως ε, κάποια επίμαχα θέματα, ιδιαίτερα όπως το θέμα της αλλαγής του κλίματος που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες λόγω της διαφορετικής θέσης των διαφορών κρατών μελών. Σίγουρα είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα πρέπει πρώτα να συζητηθεί εσωτερικά. Πολύ σημαντικό όμως είναι να υπάρχει μια βάση για τη συζήτηση διότι θα πρέπει να καθορίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος, ε, σας ευχαριστώ. Ήθελα να πω πριν ότι μετά το καλοκαίρι θα ε, έχουμε κάποιες εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλες ε, τις προκλήσεις συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προκλήσεων. Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα. Θα υπάρξει και ένα έγγραφο στρατηγική από πλευρά τη Κομισιόν σχετικά με τι θεσμικέ δυνατότητε. Είμαι βέβαιη λοιπόν ότι θα σα ε, ξαναδούμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά Έχουμε ηχογραφήσει τις παρεμβάσεις σας. Αν ε, ε, έχετε κάποια έγγραφα τα οποία πιστεύετε ότι θα είναι χρήσιμα και που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, θα θέλαμε πολύ να τα λάβουμε. Ε, ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε χρόνο για διάλειμμα.